Μία ανακοίνωση. Οι αυστριακές αρχές μου είπαν, μου ζήτησαν να αρθεί η ασυλή του Hans Peter Martin, δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2 του κανονισμού. Και αναπέμπεται αυτό το αίτημα στη Νομική Επιτροπή. Παραπέμπεται με